να βοηθήσουν στην ενίσχυση της κοινοβουλευτικής συνεργασίας καθώς και την ε, καλύτερη ε, συνεργασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Now I give the floor to our next speaker. Επόμενος ομιλητής η κυρία Φαν Μπρέμπτ. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ακούγοντας κανείς τη σημερινή συζήτηση διαπιστώνει το εξή. Ε, όλες οι πολιτικές ομάδες σχεδόν ζητούν οικονομική διακυβέρνηση. Είναι φαινομενική αυτή η ομοφωνία γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά στον τρόπο με τον οποίο αυτό το ερμηνεύουμε. Ε, το Συμβούλιο για παράδειγμα, το είδαμε αυτό και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, ε, μιλάει για μια μονομερή εστίαση σε αυτά που θεωρεί το Συμβούλιο σκόπιμα. Δηλαδή, ε, περικοπές, περικοπές, περικοπές τι κάνουν την ε, ιδεολογία τους ε, οικονομική νομοτέλεια ότι αρκεί να κάνεις μεγάλες οικονομίες και όλα θα πάνε καλά αυτό δεν είναι η δική μας ερμηνεία της οικονομικής διακυβέρνησης άλλο πράγμα χρειάζεται, πολύ διαφορετικό και δεν το λέμε μόνο εμείς αυτό ρωτήστε και οικονομολόγους και τους χτεσινούς Financial Times που δεν είναι και σοσιαλιστικό ε, όργανο προπαγάνδας λέει όταν γίνονται τόσες πολλές περικοπές και τόσες οικονομίες ε, οι οικονομίες αυτές ε, αδυνατίζουν και είναι όλο πιο δύσκολο να πληρώσουν τα χρέη τους τελικά. Αυτό που χρειάζεται είναι και επενδύσεις. Ωραίο παράδειγμα και πρακτικό να σας φέρω ε, ας πούμε, πώς θα αυξηθεί η απασχόληση. Αν υπάρχουν περισσότερες θέσεις εργασίας, τότε θα μπορέσουν τα κράτη να πληρώσουν τα χρέη τους. Εκεί θα πρέπει να επενδύσουμε λοιπόν στην εργασία ε, και να αφήσουμε αυτές τις περικοπές. Γιατί δεν πρόκειται να μας οδηγήσουν σε αυτή ε, τη λύση. Χρειάζεται και όραμα οικονομικό. Και μετά τους απαραίτητους πόρους να βρούμε για να το ελοποιήσουμε. Τώρα έχουμε το σύμφωνο σταθερότητα, αλλά προ αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να το ε, κατευθύνουμε, να το στρίψουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ράντζελ, για 1,5 λεπτό επίση. Πρόεδρε, Κύριε Πρόεδρε του, Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήθελα και εγώ να πω ότι η θέση του ΕΛΚ είναι σαφής Πιστεύουμε ότι η επίλυση της κρίσης αυτής, της οξύτατης κρίσης που περνάει η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βρεθεί μόνο εάν έχουμε περισσότερη οικονομική συνεργασία και κοινοτικό σύστημα. Για μας ε, κοινοτική μέθοδο μάλλον. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι χωρίς την κοινοτική μέθοδο, χωρί την οικονομική διακυβέρνηση, χωρί τα ίδια τα εργαλεία ενός ενιαίου νομίσματος που να είναι αληθινό στο χώρο της Ευρωζώνης δεν υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπίσουμε και να διορθώσουμε τα προβλήματα της κρίσης. Αυτό σημαίνει όμως ότι κάθε ένα από τα θεσμικά όργανα, το Συμβούλιο, η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αναλάβουν πλήρως τις ευθύνες τους έναντι των πολιτών είναι σημαντικό να γίνει εδώ σαφές ότι τα μεγαλύτερα κέρδη του, Ευρω η πιο αποτελεσματικοί μέθοδοι του Κοινοβουλίου μπορούν να τεθούν στην υπηρεσία τη κοινοτική μεθόδου προκειμένου να ενισχύσουμε το ιερό νόμισμα και την οικονομική διακυβέρνηση και να έχουμε τι απαραίτητε προποθέσει για να βοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να βγει από αυτή την κρίση. Και είναι επίση προφανέ ότι σήμερα ο ίδιο ο χώρο τη Ευρώπη, όπω μα είπαν ε, ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αντίκεινται σε όσα είπε η κυρία Φεραίρα και οι σοσιαλιστέ. Θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν με έργαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά προ όφελο των Ευρωπαίων πολιτών. Θα πρέπει όλοι να λάβουμε τι ευθύνε μα, και το Συμβούλιο και η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Και αυτό ήθελα να επισημάνω και στον πρόεδρο τη Επιτροπή, τον κύριο Μπαρόζο, και του Συμβουλίου, τον κύριο, τον κύριο Φανρόμποη. Ευχαριστούμε. Η κυρία Γιαννάκου, για ένα μισή λεπτό. Είναι προφανές ότι ο μόνιμος μηχανισμός στήριξης που αποφασίστηκε είναι οπωσδήποτε θετικό βήμα. ωστόσο λείπει ακόμα ο στρατηγικός σχεδιασμός που θα έπρεπε να περιλαμβάνει την οικονομική ένωση και προφανώς την οικονομική διακυβέρνηση. η ευρωπαϊκή ένωση δημιουργήθηκε χάρη στις ισχυρές κυβερνήσεις της εποχής. η οικονομική κρίση μπόρεσε να περάσει χάρη σε αδύναμες κυβερνήσεις που επέτρεψαν στους οικονομικούς αυτοματισμούς της οικονομικής παγκοσμιοποίησης να υποκαταστήσουν τις πολιτικές αποφάσεις που η κοινωνία μας έχει ανάγκη για να διατηρήσει τη λειτουργία της. η ευρώπη εξασφάλισε 50 χρόνια ευημερίας και εμείς σήμερα είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε να εξασφαλίζουμε αυτή την ευημερία στους πολίτες. είναι σαφές λοιπόν ότι πρέπει η ανάπτυξη να συνεχιστεί. το ερώτημα είναι ποια είναι η ανάπτυξη σε μια εποχή που όλα αλλάζουν στο παγκόσμιο σύστημα. τι είναι η ευρώπη τι θα είναι χώρα βιομηχανιών μικρομεσαίων επιχειρήσεων υπηρεσιών εξαγωγικός παράγων. χρειαζόμαστε λοιπόν ισχυρότερη ευρώπη αντί για την καχυποψία και τον διακυβερνητισμό που εμφανίζονται πολύ συχνά τελευταία. είναι ολοφάνερο ότι ορισμένε χώρε δεν τήρησαν το σύμφωνο σταθερότητα αλλά όπω ο κύριο ράινφελντ πέρσι το δεκέμβρη μου απήντησε μόνο μία χώρα τήρησε πλήρω το σύμφωνο σταθερότητα. όλε οι άλλε δεν τήρησαν τι υποσχέσει τους επομένως θα πρέπει να στηρίξουμε όλοι μαζί τις χώρες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη δίνη της κρίσης γιατί σε τελευταία ανάλυση πού βρίσκεται η δύναμη των μεγάλων χωρών; νομίζω στην κοινή παρουσία των μικρών χωρών μέσα στο ευρωπαϊκό σύστημα. άλλωστε το κόστος της μη ευρώπης κύριε πρόεδρε είναι οπωσδήποτε δυσβάστακτο για όλους μας. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Κέλαμ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, συνάδελφοι. Το κλειδί για να ξεπεράσουμε την οικονομική κρίση είναι να καταλήξουμε σε ορισμένα συμπεράσματα από αυτή, διότι πρόκειται για κρίση εμπιστοσύνης και ευθύνης, καταρχήν. Η εμπιστοσύνη αφορά έχει σχέση με λογικές δαπάνες και η Ευρώπη είχε μάθει να καταναλώνει σε βάρος του αύριο και του μεθαύριο, σε βάρος της επόμενης γενιάς, των οποίων οι αριθμοί μειώνονται δραματικά. Δεύτερον, έχουμε συνηθίσει ε, ε, να κάνουμε ορισμένα πράγματα και έχουμε διαπιστώσει ότι ορισμένοι ακολουθούν το, έχουν την τάση να ακολουθούν το παράδειγμα των μεγάλων χωρών. Η αρχή της δημοσιονομικής πειθαρχίας πρέπει, πρέπει να εφαρμόζεται με μεγαλύτερη αυστηρότητα από αυτό θα κριθεί η αξιοπιστία της Ευρώπης. Τρίτον, υπάρχει ανάγκη για μηχανισμούς εξασφάλισης ισορροπιών. Δεν μπορώ παρά να εγκρίνω τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την οικονομική διακυβέρνηση, την ενεργοποίηση των κριτηρίων για το χρέος και τη δυνατότητα για έναν ε, ε, μηχανισμό έγκαιρης παρέμβασης και υποστηρίζω τα συμπεράσματα του συναδέλφου Φερχόφσταφ. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ουσιαστική οικονομική διακυβέρνηση και ένα σύστημα αυτόματων κυρώσεων προσβλέπουμε στο προτάσεις πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μελλοντικό μηχανισμό ε, επίλυσης της κρίσης τον επόμενο μήνα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Κέλλαμ. Πάμε τώρα στη διαδικασία Catch the Eye και θα δώσω το πρώτο το λόγο στην κυρία Μπασέσκου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να καλωσορίσω τη λήψη νέας δέσμης μέτρων για την ενίσχυση της δημοσιονομικής ε, πειθαρχία και την επέκταση της οικονομικής παρακολούθησης. Πραγματικά όλα αυτά είναι απαραίτητα γιατί είδαμε διαφορές στα κράτη-μέλη ε, με το τι πολιτικές ακολουθούν και πόσο σέβονται τον προπολογισμό τους. Η οικονομική κρίση ε, οδήγησε σε ανησυχητικές σε διάφορες χώρες και μεταξύ των χωρών αυτών είναι και η Ρουμανία. Θεωρώ ότι αυτό που χρειάζεται είναι ένα νέο πλαίσιο μακροοικονομικής επαγρύπνησης για να μπορούμε από νωρί να ανοιχνεύουμε τους κινδύνους και τις ανισορροπίες. Η οικονομική διακυβέρνηση και η πρόταση της ομάδας εργασίας του κυρίου Βαν Ρομπεϊ είναι ένα βήμα προς τα εμπρός, απομένει να εφαρμοστεί για να δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο διαχείρισης κρίσεων. Κατά τον ίδιο τρόπο θα ήθελα να αναφέρω πόσο σημαντικό ε, θεωρώ το θέμα του κανονισμού ε, που παρακολουθεί ε, τους προπολογισμού των κρατών μελών. Στο μέλλον κανένα κράτος δεν θα μπορεί να παραβιάζει τα κριτήρια αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Προεδρία, η Ουγγρική, ε, θα έχει να αντιμετωπίσει μια ε, τεράστια πρόκληση. Αναθεώρηση της συνθήκης της Λισαβόνας και οικονομική διακυβέρνηση. Πολύ μεγάλη πρόκληση, επαναλαμβάνω. Ε, τα νέα κράτη-μέλη εκτός της Ευρωζώνης παρακολουθούν με πολύ μεγάλη αγωνία τα τεκτενόμενα εντός της Ευρωζώνης. Βεβαίως θα πρέπει να έρθουμε πιο κοντά στην Ευρωζώνη και εμεί, αλλά για να γίνει αυτό έχουμε υποχρεώσεις. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και πρέπει να σας πω ότι αυτά που τώρα συμβαίνουν στην Ιρλανδία μας ανησυχούν πάρα πολύ γιατί έπονται δεχομένω και η Πορτογαλία και η Ισπανία. Πολλοί μας έχουν θορυβήσει. Δεν μπορεί να καταρρεύσει η Ευρωζώνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδρασε αργά με αν μη τι άλλο πήρε τη σωστή απόφαση. Και πραγματικά θα είναι σταθμός στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ναι, στην οικονομική διακυβέρνηση βεβαίως οπωσδήποτε. Υπάρχουν όμως ακόμα πολλά εμπόδια όπως γνωρίζουμε. Εγώ πιστεύω ότι η Ουγγρική Προεδρία θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι τη για να βοηθήσει την κατάσταση. Ευχαριστώ. Η κυρία Φιγκερέιντο, παρακαλώ. Η μεγαλύτερη γενική απεργία των τελευταίων 20 χρόνων αυτός ο αγώνας και άλλες πολύ σημαντικές σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Ελλάδα ή η Γαλλία δείχνουν ότι απαιτείται απόκριση από του βασικού υπεύθυνου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ποια είναι αυτή, αγνοούν τι διαμαρτυρίε με τι αντικοινωνικέ του πολιτικέ και επιμένουν στι ίδιε πολιτικέ που συνέβαλαν στην κατάσταση στην οποία έχουμε οδηγηθεί. Αυτό σημαίνει ότι το να είναι ευάλωτο το ευρώ είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο προκύπτει τι πολιτικέ που επικρίνονται, την απελευθέρωση του αγορά κεφαλαίων και την οικονομική κερδοσκοπία χωρί όρια. Οι απαιτήσει για την ονομαστική ε, λογοδοσία μέσω του ε, Συμφώνου σταθερότητα χωρί την πραγματική σύγκληση των οικονομιών βλέπουμε ότι επιδιώνονται η ανεργία και η ένδυα που έχουν φτάσει σε επίπεδα ανυπόφορα και οι κοινωνικέ πραγματικότητε όλο ένα υποβαθμίζονται. Τι θα γίνει λοιπόν με αυτή την κατάσταση, τι θα κάνουμε για το ευρώ, Πώ θα επιμένουμε σε αυτέ τι πολιτικέ και θα επιμένουμε πάντοτε στην παραγωγή την, ε, χωρίς να, δίνουμε καλύτερη θέση στην ε, εργασία και την απασχόληση. Ε, κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έλαβε χώρα στα τέλη Οκτωβρίου και όλα τα κράτη-μέλη διορθώνουν τώρα την οικονομική πολιτική τους προκειμένου να εξασφαλίσουν κάποια ανάπτυξη μετά την Ιρλανδία και την Ελλάδα και άλλες χώρες πιθανώς να αντιμετωπίσουν δυσκολίες. Είναι λοιπόν σαφές ότι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων δύσκολα μπορούν να αποφασίσουν. τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να συζητήσουμε για το κοινό μας όραμα για να βγούμε από την κρίση το ταχύτερο δυνατό. Δεν πρέπει να υποτιμούμε τις προσπάθειες των κυβερνητικών εκπροσώπων. Και βεβαίως πρέπει να λάβουμε υπόψη τα συμφέροντα της Ευρώπης. Ο κύριος Μπρόντς. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει ότι πρέπει να αποφύγουμε κάθε μορφή προστατευτισμού και κοιναλαματικές ε, ε, κινήσεις. Η υιοθέτηση του φιλελευθερισμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε ε, θύματα τις χώρες από τις αναδυόμενες οικονομίες, στην Κίνα ειδικότερα, με την οποία δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε. Υπάρχει πρόβλημα με το copyright, απασχολούν εργαζόμενους με γελίους μισθούς και προσπαθούν να μειώσουν ακόμα περισσότερο τις αμοιβέ. Πρέπει ε, ε, να προστατεύσουμε τις επιχειρήσεις και τους υπαλλήλους από αυτό τον αθέμητο ανταγωνισμό. Για... Δεν πρέπει να διατηρου... πρέπει να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε σε λογικά επίπεδα το ευρώ. Εάν το νόμισμα ορισμένων χωρών υποτιμάται, θα ακολουθήσουν και άλλα αυτή την πορεία. Ευχαριστώ κύριε Μπρόντς και θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Πρόντι. Οντί. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύω. Ε μάλλον κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου και Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, τι δεν γίνεται με τις δημόσιες δαπάνες στην Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε μεγάλες προκλήσεις. Δεν θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε με τους εθνικούς βουλευτές, τους συναδέλφους και φίλους, το θέμα της κινητικοποίησης, δηλαδή ε, ε, της ε, αμοιβαίας υποστήριξης. Ε, ε, το είπε και ο Λαμασούρ, γιατί να έχουμε 25, 27 στρατούς χωρίς εχθρό, γιατί να έχουμε διάφορες φορολογικές ας πούμε, ε, υπηρεσίες διαφορετικές, δεν μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας στην ενέργεια, στις μεταφορές και αλλού. Δεν μπορούμε να θέσουμε σε ένα εξωτερικό ε, οικονομικό ελεγκτή να κάνει τον έλεγχο στα τρία επίπεδα, στο ευρωπαϊκό, στο εθνικό και στην τοπική αυτοδιοίκηση και να μας φέρουν αυτό το audit, τον οικονομικό έλεγχο και στα εθνικά κοινοβούλια και ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Ελεκτικό Συνέδριο και στα 27 Εθνικά Ελεκτικά Συνέδρια για να κάνουμε καλύτερη διαχείριση των δημοσίων δαπανών σε όλη την Ευρώπη από κοινού. Ευχαριστώ. Μπενόβα. Κυρία Φλασίκο Βαμπένοβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε της Επιτροπής, συνάδελφε. Το... Η Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ουσιαστικά ασχολήθηκε με τη συζήτηση για την οικονομική ύφεση και τις συνέπειές της. Με αυτό, γι' αυτό συζήτησαν οι αρχικοί κατόχοι κυβερνήσεων. Δεν αρκεί μόνο οικονομική διακυβέρνηση όμως, χρειάζονται και άλλες διαφορετικές αλλαγές που να ασχοληθούν απευθείας με το χρέος. Ο κάθε μηχανισμός θα πρέπει να καλύπτει όλα τα ζητήματα, πέραν του απλού χρέους όμως. Ή αποκλειστικά του χρέους. Ιδάλλως δεν θα λειτουργήσει η μεταρρύθμιση του συστήματος των συντάξεων, οι συνέπειες στα ελλείμματα, όλα αυτά έχουν αρχίσει να γίνονται ένα ζήτημα με όλα ένα μεγαλύτερες διαστάσεις ασχολούμαστε πάρα πολύ με τις λεπτομέρειες. Εάν ε, η μεταρρύθμιση των συντάξεων ήταν τόσο απαραίτητη όσο ακούγεται, θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες, γιατί δεν είναι μόνο οι συντάξεις που επιβαρύνουν τα ελλείμματα. Αυτό είναι λογικό. Και καθώς οδεύουμε προς την ιδέα συνολικών λύσεων, δεν μπορούμε συνεχώς να προβλέπουμε εξαιρέσει. Ε, thank you, ε, Mr. Ο κύριος Μπάστον, ευχαριστώ πρόεδρε. Απλώς λίγα σχόλια για όσα υπόθηκαν το πρωί από τον πρόεδρο Φαν Ρόμπεϊ και τον κύριο Μπαρόζο. Φαίνεται ότι και οι δύο αρνούνται την πραγματικότητα. Αρνούνται το γεγονό ότι η Ευρωζώνη αντιμετωπίζει κρίση και βρίσκεται στο χείλο τη καταστροφή, τη κατάρρευση. Για πολλού επίση, ακούσαμε και αυτοί να αρνούνται την πραγματικότητα. Πρέπει να ξυπνήσουν οι πολίτε υποφέρουν στις χώρες τους και καταλαβαίνουν ότι είμαστε πολλοί εδώ, πολλοί και δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη μεγαλύτερη κρίση που έχουμε ποτέ. Τα πράγματα είναι πια σοβαρά. Θέλω ο κύριος Μπαρόζο και ο κύριος Ρόμπεϊ να μου πούν παρακαλώ, ε, όσο και λίγο να μιλήσουν, ποιο είναι το πρόγραμμά τους. Πρέπει να υπάρχει μια δεύτερη επιλογή, ένα plan B. Τι θα κάνετε για αυτές τις εκλογές. Πιστεύω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη κρίση που αντιμετωπίσαμε ποτέ. Τα κράτη-μέλη πλήττονται όλα. Πάντοτε περιμένει κανεί από του πολιτικού ε, ηθήνοντε να έχουν και μια δεύτερη επιλογή, μια δεύτερη εναλλακτική. Πείτε μα ποια είναι αυτή. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκάλπελτ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σημειώνω με χαρά το γεγονό ότι η μεταρρύθμιση του συνεργατικού συστήματο κρίθηκε σημαντική από το Συμβόλιο. Υπάρχει και το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη και οι ίσε ευκαιρίε δεν παρέχονται σε όλου σύμφωνα με αυτό το σχέδιο. Έγιναν διακρίσει, έτυχε διακριτική μεταχείριση η, Πορτο... η Πολωνία. Είπαμε ότι είναι σημαντικό το θέμα τη μεταρρύθμιση του συνεργατικού συστήματο. Δεν πρέπει να γίνονται διακρίσει υπέρ κρατών μελών και να το αποφύγουμε αυτό που να λάβουμε υπόψη διαφορετικέ συνθήκε να καθορίζουμε τον προπολογισμό για τα διάφορα θέματα. Είναι ένα θέμα που πρέπει να λυθεί. Τα ευχάριστα νέα ότι έχουμε το θέμα αυτό ήδη στο ενημερήσια διάταξη του Συνόδου Κορυφή του Συμβουλίου το Δεκέμβριο και σα καλώ να πάρετε μία ε, απόφαση που δεν θα οδηγήσει σε διακρίσει. Όταν μιλάμε για νομοθεσία, νομοθετικό έργο στο μέλλον, πρέπει αυτή η διαδικασία να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό, διότι πρέπει να ολοκληρωθεί αυτό το θέμα με μια λύση που θα ικανοποιήσει όλους. Η κυρία Παπαδοπούλου. Πρόεδρε, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία βιώνουν τι συνέπειε τη οικονομική κρίση. Η ασκή του αιώλου άνοιξαν ήδη. Η λήψη μέτρων είναι πια μονόδρομο. Η καχυποψία και ο ευρωσκεπτικισμό δεν συμβάλλουν στην επανάκαμψη από τη διεθνή οικονομική κρίση. Αντίθετα, αυτό που χρειάζεται είναι κοινοτική αλληλεγγύη, πολιτική βούληση, όραμα, εμπιστοσύνη στον δυναμισμό τη Ευρώπη και πρωτίστω συντονισμένε δράσει. Δράσει για διαρθρωτικέ αλλαγέ σε επίπεδο χωρών αλλά και στην ευρωπαϊκή ένωση αύξηση τη απασχόληση, αύξηση τη ανάπτυξη, επιτάχυνση αύξηση των θέσεων εργασία, υλοποίηση της στρατηγικής Ε, ε, ε, ε Εξορθολογισμό και εξηγίαση τη εταιρικής διακυβέρνηση, διαφάνεια στην οικονομική διακυβέρνηση έλεγχο στα εθνικά στατιστικά δεδομένα μόνιμος μηχανισμός μηχανισμό διαχείριση κρίσεων ε, ε, στην ευρωπαϊκή ένωση προ όφελο πάντα του ευρωπαίου πολίτη. η κρίση αφορά όλου και όχι μεμονωμένα τι χώρε που τη βιώνουν. αυτό που απαιτείται είναι κοινοτική αλληλεγγύη και συντονισμό δράσεων. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Now, Mr. Ο κύριος Μάντλενερ τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωζώνη τώρα καταραίει και ο κύριος Μπαρόσο ε, θα πρέπει να συνοδεύει αυτή την κατάρρευση. Ε, δισεκατομμύρια δίνουμε εδώ και χρόνια σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Ισπανία αλλά δεν μπορούσαν οι οικονομίες τους να είναι ανταγωνιστικές των μεγάλων οικονομικών της Ολλανδίας ε, και της Γερμανίας. Βλέπουμε πού οδηγεί η πολιτική των ε, σοσιαλιστών. Στην Ελλάδα το 1 τρίτο του πληθυσμού σχεδόν είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Και βλέπουμε τι γίνεται και με τη μετανάστευση, τσουνάμι ε, και είναι και άνεργοι και έχουν εγκατασταθεί στις χώρες μας. Η Ισπανία ένα εκατομμύριο λαθρομετανάστες τους νομιμοποίησε και έχει ξεπεράσει η ανεργία της το 20%. Πάλι δισεκατομμύρια θα τους στείλουμε. Δεν είναι πολύ ακριβό αυτό βραχυπρόθεσμα Μάκρο μακροπρόθεσμα θα τεθεί το ερώτημα. Είμαστε διατεθειμένοι ε, ε, να συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε αυτές τις ασθενείς χώρες με χρήματα των δικών μας φορολογουμένων. Η απάντηση είναι όχι. Μήπως να ξαναφέρουν τη δραχμή στην Ελλάδα ή το παλιό τους ε, νόμισμα τη λίρα στην Ιρλανδία για να λύσουμε τα προβλήματα. Και να τα συζητήσουμε αυτά τα θέματα σοβαρά με τις ενδιαφερόμενες χώρες. Ευχαριστώ κύριο Σκέλη. Ω Ιρλανδό βουλευτή, καθόλου δεν χαίρομαι να βρίσκομαι εδώ σήμερα και να ακούσω όλου του ομιλητέ να αναφέρονται στην Ιρλανδία λόγω τη οικονομική μα κατάσταση. Ιδιαιτέρω, γιατί πριν από λίγα χρόνια ήμασταν σχεδόν ένα οικονομικό παράδειγμα για την Ευρώπη, για την επιτυχία μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ε, έχει ληφθεί απόφαση στην Ιρλανδία να διορθώσουμε τα πράγματα και ο λαό τη Ιρλανδία καλωσορίζει την βοήθεια από του Ευρωπαίου φίλου και συναδέλφου. Είναι αρκετά τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει από αυτή την εμπειρία. Ε, ε, πολλοί μίλησαν για χαζομάρα και απληστία των Ιρλανδών πολιτικών που ήταν μέρο του καπιταλιστικού συστήματο που έδινε ωφέλη στι τράπεζες και τους ρυθμιστέ. Ε, όμως ε, το ρυθμιστικό οικοδόμημα που θα προκύψει από το ε, κουτί εργαλείων του πακέτου οικονομικής διακυβέρνησης είναι κάτι που θα μας βοηθήσει στο μέλλον να παρακολουθούμε το τι συμβαίνει και να τους ανακαλούμε στην τάξη όσους περνούν σε παρασπονδίες. Ευχαριστούμε κύριος Μπαλσίτης. Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, Σήμερα αρχίσαμε να μιλάμε για πολύ σημαντικά θέματα. Το θέμα της μελλοντική οικονομικής διακυβέρνησης ειδικότερα και σύντομα επίσης θα συζητήσουμε για, την, για ένα κοινό σύστημα φορολόγησης. Εφόσον βλέπουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις πάνω στην οικονομία μας ενός ισχυρού ευρώ ε, Έγινε το τεστ αντοχή των τραπεζών πριν από έξι μήνες και τα αποτελέσματα αποδείχθηκαν απογοητευτικά. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε αξιόπιστα στοιχεία, αξιόπιστες πληροφορίε. Δεν θα μπορέσουμε λοιπόν να ξεφύγουμε εύκολα από αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Καλό λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δραστηριοποιηθεί περισσότερο σε ό,τι αφορά την υποβολή νομοθετικών προτάσεων στο μέλλον, διότι θα χρειαστούμε περισσότερες προσπάθειες, μεγαλύτερη κινητοποίηση και αυστηρότερους ελέγχους οικονομικούς και άλλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Βέρ. Ε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, λαμβάνω σύντομα το λόγο στη συζήτηση αυτή. Έχουμε καταλάβει πλέον ποιος φταίει για την κρίση. Ένα τμήμα του τραπεζικού τομέα που έκανε ακάλυπτες, πολύ ε, ρηψοκίνδυνες συναλλαγές και κυβερνήσεις που δεν είχαν ε, υπόψη τους τις οικονομίες που έπρεπε να κάνουν και τη χρηστή διαχείριση του προπολογισμού. Ε, χρειάζεται τώρα όσο γίνεται μεγαλύτερη αλληλεγγύη για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, λένε ορισμένοι, ενώ ε, άλλοι ζητούν μεγαλύτερη ευθύνη για να βγούμε από την κρίση. Δεν θα ήταν σωστό, πιστεύω, να μην πληρώσουν την κρίση εκείνοι οι οποίοι ευθύνονται για την κρίση. Αυτό που χρειάζεται τώρα δεν είναι περικοπές ε, προς πάσα κατεύθυνση. Θα πρέπει ε, να βοηθηθούν οι χώρες... Α, ο πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή, τελείωσε ο χρόνος. Ευχαριστώ. Ο Πετρουλούχαν. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Η έκθεση για την οικονομική διακυβέρνηση είναι ένα σημείο θετηρίας. Θα πρέπει να εξεύρουμε ένα σύστημα βιώσιμο ε, για να λειτουργήσουν όλα αυτά. Οι συστάσεις της έκθεσης ε, για ισχυρότερα θεσμικά όργανα, για αποτελεσματικότερη οικονομική διακυβέρνηση, οι συστάσεις που αφορούν τη δημιουργία σε επίπεδο διακρατικό τέτοιων ε, φορέων που να μπορούν να δώσουν αξιολογήσεις ανεξάρτητες, αποτιμήσεις και προβλέψει για φορολογικά ζητήματα είναι τα απαραίτητα θεμέλια για να έχουμε ένα σύστημα διαφανέ που να λειτουργεί για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι θα πρέπει κάθε κράτο μέλο να έχει τη δυνατότητα να εξηγήσει με σαφήνεια ποια είναι η βάση της ανάλυσης του για κάθε φορολογικό μέτρο που θα προτείνει χρειαζόμαστε μια προσέγγιση που να βασιστεί στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και την αμοιβαία αναγνώριση. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένα στοχευμένα μέτρα που θα μας επιτρέψουν να έχουμε οικονομική διακυβέρνηση αξιόπιστη, διαφανή, κατά τρόπον ώστε να μπορεί να γίνει συζήτηση για οποιοδήποτε μέτρο υιοθετείται σε οποιοδήποτε κάτω μέλο. Μέτρα τα οποία στη συνέχεια μπορεί να έχουν συνέπειε στο σύνολο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε. Έχουμε δύο ακόμη αγορητέ. Πρωτού δώσω το λόγο στον πρόεδρο Μπαρόζο. Η κυρία Φερέιρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να Ζήτησα ξανά το λόγο γιατί είχα ζητήσει προηγουμένως να παρέμβω ε, με τον ε, κανόνα της γαλάζιας κάρτας. Διότι με ανέφερε ο συνάδελφο Ραντζέλ. Ε, ήθελα λοιπόν ε, να μου είχατε δώσει νωρίτερα το λόγο για να, για να απαντήσω. Τέλο πάντων, εποφελούμε για να πω στον συνάδελφο Ραντζέλ ότι καλό θα να μα εξηγήσει σε όλου ποια είναι η άποψή του για τι πραγματικέ ε, διαφορές των όσων των προτάσεων τη ε, καγκελαρίου Μέρκελ και των προτάσεων τη Επιτροπή σε σχέση με το δημόσιο χρέο. Ήθελα να μα το πει αυτό. Διότι η πρώτη πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πραγματικότητα ήταν ευρωπαϊκή. Οι προτάσει για το δημόσιο χρέο όμω πήγαν στον κάλαθο των αχρήστων. Ε, και παρόλη την δημόσια συζήτηση που έγινε. Τι έγινε λοιπόν με την εξυπηρέτηση των συμφερόντων τη Γερμανία. Obrigado. Ευχαριστώ. Κύριε Ράντζελ, Θέλετε να απαντήσετε. Πολύ σύντομα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι στην ευρωπαϊκή διαδικασία Προφανώ υπάρχουν διαρκεί διαπραγματεύσει μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Όμω η θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμόνως ε, υποστήριζε την κοινοτική προσέγγιση και την ε, ισχύ του ενιαίου νομίσματος. Ξέρω ότι κάποιοι βουλευτές θέλουν να κάνουν εθνική πολιτική στο πλαίσιο του Ευρωκοινοβουλίου και αυτή είναι και περίπτωση της κυρίας Φερέιρα. Thank you. Ευχαριστούμε. Και τέλος, σε αυτό το γύρο, ο κύριος Φιέλ. Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια περίοδο μεταρρυθμίσεων Απαιτείται λοιπόν απόκριση στην κρίση και απαιτείται και υπεράσπιση του ενιαίου νομίσματος. Ένα νόμισμα που χρειάζεται κανόνες ενιαίους κοινού που να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα μέλη. Το Ευρωκοινοβούλιο ήδη έχει τοποθετηθεί μια, σε μια πρώτη φάση σε ό,τι αφορά την οικονομική διακυβέρνηση. Ε, και είναι υπέρ μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων κρατών σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και τη σταθερή ε, και αποφασιστική υλοποίηση του Συμφώνου Σταθερότητα. ώστε να υπάρχει συντονισμό μεταξύ των κρατών. Και θα πρέπει να είναι το πρώτο θεσμικό όργανο το Ευρωκοινοβούλιο που θα ε, ασχοληθεί με την κατάρτιση, την ίδρυση ενό ταμείου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του δημοσίου χρέου των κρατών έτσι θα πρέπει να συνεχιστεί η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, συγχαίρουμε για τον έργο του τον Πρόεδρό τη και επίση σκοπεύουμε να συνεχίσουμε και τη συνεργασία μα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σε αυτήν την ε, διαδικασία έχουμε τόσε εκθέσει που έχουν συζητηθεί και η τοποθέτησή μα πλέον έχει γίνει σαφή. Ευχαριστούμε. Τώρα, συνάδελφοι, προκειμένου να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μα και να απαντήσετε και κάποιε ερωτήσει, να δώσω το λόγο στον πρόεδρο Μπαρόζο. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Αγαπητά μέλη, αξιότιμοι βουλευτές, θα απαντήσω σε ορισμένες συγκεκριμένες ερωτήσεις και μετά θα προβώ σε συγκεκριμένα σχόλια. Το θέμα που έθιξε ο κύριος Σούλς καταρχήν, άκρο σημαντικό, για τα τεστ αντοχής της Ιρλανδίας. Η κοινή μεθοδολογία συμφωνήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, και πρόκειται για μια αυστηρή διαδικασία με μακροοικονομικά σενάρια. Στη συνέχεια, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, εποπτικές αρχές έπρεπε να αναλάβουν την εκτέλεση αυτή. Όπως όρισε και η ΕΚΤ, δεν υπήρχαν ευρωπαϊκές αρμοδιότητες επ' αυτού. Και μέχρι πρόσφατα δεν μπορούσαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να φέρουμε τέτοια ευθύνη. Αυτό βεβαίως θα αλλάξει στο μέλλον. Θα έχουμε το νέο οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής και Ρυθμιστικής Αρχής μετά από συμφωνία του Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα υπάρχει προληπτική εποπτεία και ένα ασφαλιστικό ε, σύστημα καθώς και ένας χρηματοοικονομικός εποπτικός μηχανισμός. Και έτσι θα έχουμε καλύτερους μηχανισμούς και υποδομή έτσι ώστε να γίνουν αυτές οι δοκιμές αντοχής στο μέλλον κατά πιο σαφή τρόπο και αποτελεσματικό. Άρα πριν από την κρίση δεν είχαμε στη διάθεσή μας τα μέσα που διαθέτουμε τώρα. Και τώρα φτάνω στο δεύτερο θέμα, το θέμα του πώς αντιμετωπίζουμε ορισμένα επίμαχα θέματα όπως το μηχανισμό μονίμων κρίσεων. Το μόνιμο μηχανισμό κρίσεων, με συγχωρείτε. Θα ήθελα να τονίσω ότι ομόφωνα οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αποφάσισαν να ζητήσουν τη σύσταση ενός μόνιμου μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων. Εγώ τόνισα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τους ε, ενεχόμενους κινδύνους τη στιγμή που δεν θα υπήρχε η σωστή προετοιμασία. Το θέμα όμως εφήγει και θα πρέπει τώρα να το αντιμετωπίσουμε κατά αποτελεσματικό τρόπο. Γι' αυτό και ακούστηκαν ε, ορισμένα σχόλια τα οποία δεν βοηθούν καθόλου την κατάσταση. Αντιμετωπίζουμε μία δύσκολη, μία δυσχερή κατάσταση. Τώρα χρειαζόμαστε δράση και όχι σχόλια. Έχουμε να κάνουμε με ιδιαίτερα ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν το παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα. Νομίζω λοιπόν ότι δεν μας βοηθάει να μιλάμε απλώς για κινδύνους. Θα πρέπει να προετοιμάσουμε όλους τους μηχανισμούς έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια χρηματοοικονομική και δημοσιονομική σταθερότητα. Γι' αυτό δεν θα μιλήσω για σχέδιο Β αυτό τόνισε και ο πρόεδρος Βαν Ρόμποϊ. Τονίζουμε και συζητάμε αυτά τα ζητήματα μέσα στα πλαίσια κοινή ευθύνη με τα κράτη-μέλη. Η Επιτροπή πάντα προωθούσε φιλόδοξα προγράμματα. Είμαστε υπέρ μιας φιλόδοξης οικονομικής διακυβέρνησης για την Ευρώπη. Όμως θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Δεν μπορούμε να κινηθούμε πέραν των κοινών συμφωνιών από τα κράτη-μέλη. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Όταν υφίσταται μία συμφωνία η οποία αποτελεί πρόοδο σε σχέση με την προγενέστερη κατάσταση, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ιδεώδεις καταστάσεις και μέτρα τα οποία δεν μπορούν να ισχύσουν. Εμείς λοιπόν ζητούμε να τεθούν σε εφαρμογή φιλόδοξα σχέδια αλλά και ρεαλιστικά σε σχέση με την σταθερότητα της Ευρωζώνης. Και θα ήθελα να τονίσω και κάτι άλλο. Ορισμένοι ε, μίλησαν για την Ευρωζώνη. Η Ευρωζώνη δεν ήταν το αποκλειστικό πρόβλημα. Είμαι πεπισμένος ότι η κατάσταση θα ήταν πολύ χειρότερη αν δεν υπήρχε το ευρώ. Πολύ το ξεχνάτε πολύ ξεχνάτε ότι ορισμένες χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη αντιμετωπίζουν παρόμοια και ίσως και χειρότερα προβλήματα. Και χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως η Ισλανδία, η Ισλανδία πτώχευσε και δεν διαθέτει το ευρώ. Άρα το ευρώ δεν ήταν το αίτιο του προβλήματος και από πολιτικής πλευράς είναι ανέντιμο να τονίζετε ότι το πρόβλημα έγκυται στην Ευρωζώνη. Άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να αναγνωρίσουμε τις ιδιαιτερότητες της Ευρωζώνης και να ζητήσουμε από όλα τα κράτη-μέλη μία δέσμευση έτσι ώστε να εργαστούμε από κοινού. Αυτό αφορά και όσους ανήκουν στην Ευρωζώνη και όσους δεν ανήκουν. Έτσι ώστε να υπάρχει μία κοινή αντιμετώπιση επίλυσης του ζητήματος αυτού μέσα στα πλαίσια ενός φιλόδοξου σχεδιασμού αλλά και μιας θεμητής συνεργασίας μεταξύ ενδοκινοτικών οργάνων. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θα πρέπει να αποστείλουμε. Τη στιγμή που οι αγορές κλειδονίζονται θα πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι και υπεύθυνοι μέσα στα πλαίσια ενός κοινού ευρωπαϊκού πολιτικού προγράμματος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Πρόεδρε Μπαρόζο. Τέλος, το λόγο έχει ο Πρόεδρος Βαν Ρομπόη. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Προηγουμένως είπαμε ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ανάλυση του Προέδρου της Επιτροπής και τη δική μου. Είναι η πρώτη φορά κύριε Σούτς που με κατηγορούν ότι λέω όλα πάνε καλά, αγαπητή κυρία Μαρκησία. Ζούμε ώρες δύσκολες και μόνο αν πάρετε τα λόγια μου εκτός περιεχομένου θα πείτε ότι δεν είμαι επιφυλακτικός αν. Δεν μπορεί να μιλάμε με τρόπο έντονο στο ευρωπαϊκό πεδίο. Είναι η στιγμή που πρέπει να είμαστε ήρεμοι και όχι να επαναλαμβάνουμε το βάθος της κρίσης. Το γνωρίζουμε αρκετά. Η στιγμή είναι κατάλληλη για να δράσουμε. Κύριοι, κάποιοι από εσά είπατε ότι πρέπει να πάρουμε ένα μάθημα. Στα γαλλικά λέμε ότι οι πράξεις μας μας ακολουθούν. Όταν ανέλαβα τη θέση αυτή κυρίες και κύριοι υπήρχε ένα σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης που μπόρεσε να γίνει λίγο πιο ευέλικτο πριν από μερικά χρόνια και το οποίο δεν εφαρμόστηκε. Όταν ανέλαβα κληρονόμησα τη συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία προβλέπει κάποιες διαδικασίες, μεταξύ των οποίων αφορούν, κάποιες που αφορούν ποινές, κάποιες που αφορούν ε, τις διαδικασίες που πρέπει να ληφθούν, και αυτή είναι απόφαση από, του Συμβουλίου, ε, για μια χώρα η οποία έχει υπερβολικό έλλειμμα. Όταν εγώ ανέλαβα δεν υπήρχε μηχανισμός κρίσης. Όλα αυτά χρειάστηκε να τα επανορθώσουμε, να ενισχύσουμε το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης και για πρώτη φορά να εισάγουμε ένα σύστημα μακροοικονομικής παρακολούθησης. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αν εδώ και λίγα χρόνια είχε υπάρξει αυτός ο μηχανισμός, τα προβλήματα που εμφανίστηκαν σε κάποιες χώρες ποτέ μα ποτέ δεν θα είχαν εμφανιστεί. Ανακαλύπ, ανακαλύψαμε τις φούσκες των, της, της ακίνητης περιουσίας. Ανακαλύψαμε ένα σωρό πράγματα. Τώρα έχουμε να προσθέσουμε μια κοινοτομία. ότι μαθαίνουμε πλήρως από αυτή την κρίση. Και όσον αφορά τη συνθήκη της Λισαβόνας θα την αλλάξουμε σκοπεύουμε να το κάνουμε αυτό ώστε να αποκτηθεί μια νομική βάση απέναντι σε κάποια συνταγματικά δικαστήρια μια νομική βάση για έναν μηχανισ, μόνιμο μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσης. Αυτό. Και ελπίζω ότι δεν θα μπούμε στο ρηψοκίνδυνη πορεία να αρχίσει μια μεγάλη συζήτηση για τα θεσμικά όργανα που δεν προκύπτει από πουθενά και η οποία θα αφαιρέσει ακόμα περισσότερο από την προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Δεν υπάρχουν μηχανισμοί κρίσης. Δεν υπήρξαν. Όταν αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα της Ελλάδας, χρειάστηκε να εφεύρουμε ένα μηχανισμό. Δεν υπήρχε τότε. Όταν πήραμε το άλλο μέτρο των 750 δισεκατομμυρίων της κρίσης χρειάστηκε να ερμηνευθεί δημιουργικά η συνθήκη της Λισαβόνας για να μπορέσει να στηθεί αυτός ο μηχανισμός. Αυτή τη στιγμή λοιπόν μαθαίνουμε από τις εμπειρίες μας, παίρνουμε ένα μάθημα από την κρίση και όπως λέω οι πράξεις μας θα μας ακολουθούν υπήρχε ένα σύμφωνο σταθερότητας αδύναμο που δεν εφαρμαζόταν, δεν είχαμε τίποτα για την μακροοικονομική παρακολούθηση, δεν υπήρχε μηχανισμός κρίσης. Τώρα τα κράτη-μέλη ανέλαβαν τις ευθύνες τους. Πολλά από αυτά τις ανέλαβαν. Δεσμεύτηκαν πολύ συχνά σε πολιτικές μεταρρύθμισεις που αντιβαίνουν τις μεγάλες, ε, τάσεις της κοινή γνώμης και παίρνουν πολύ συχνά εξαιρετικά θαραλέα μέτρα. Και όχι μόνο σε χώρες που υπάρχουν εντάσεις, αλλά και σε άλλες χώρες. Αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας μην κάνουμε πάντα λάθος για το ποιος είναι ο εχθρός. Γιατί υπάρχει η τάση να στρεφόμαστε όλος ιδιαιτέρως κατά των κυβερνήσεων. Μην κάνουμε λάθος. Σήμερα το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι που μιλάνε όχι μόνο για την Ιρλανδία αλλά και για την Πορτογαλία, επιτρέψτε μου να αναφέρω κάποια στοιχεία. Το κρατικό έλλειμμα 9,3 το 2009, το 10 θα είναι 7,3, 4,6 το 11. Το χρέος, το δημόσιο χρέος της Πορτογαλίας το επιτόκιο είναι κατά μέσο όρο 3,6%. Εξαιρετικά χαμηλό. Δεν πάσχει, δεν υπάρχει κρίση ακινήτων, δεν υπάρχει φούσκα ακινήτων. Ο, οικονομικός, ο χρηματοοικονομικός τομέας δεν είναι υπερβολικά διονγκωμένος σε σχέση με τη χώρα. Τα κεφάλαια των τραπεζών επαρκούν. Μην κάνουμε λάθος. Κάποιοι λένε ότι υπάρχει μια μεταδοτική τάση. Αυτή δεν στηρίζεται σε οικονομικά στοιχεία, δεν, δεν στηρίζεται στη λογική. Ας μην κάνουμε λάθος, ας μην στοχεύουμε σε λάθος εχθρό. Αυτό όσον αφορά δε, την συνεργασία μεταξύ θεσμικών οργάνων πρέπει να σας πω το εξής. Ότι σε επίπεδο προεδρίας κάνουμε τα πάντα για να, για να υπάρξει συνεργασία Δημιουργήθηκε η Task Force, ε, εγκρίθηκε από τα μέλη και τα υπεύθυνα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε άλλους τομείς του, του, μόνιμου μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων δουλεύουμε, προχωράμε χέρι με χέρι και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την κατάσταση εν ώψη του ε, προϋπολογισμού του 2011 και λοιπά που δεν υπήρξε συμφωνία. Θέλω να πω και κάτι άλλο όμως. Είστε όλοι ευρωβουλευτές, ανήκετε όλοι σε κάποιες πολιτικές οικογένειες. Οφείλω να διαπιστώσω ότι κάποιες στιγμές υπάρχει μεγάλη διάσταση ανάμεσα σε αυτά τα οποία ακούω στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από τους πρωθυπουργούς που ανήκουν σε διαφορετικά κόμματα και σε αυτά τα οποία ακούω εδώ, σε αυτό σε αυτή την αίθουσα από τα ίδια μέλη των ίδιων πολιτικών οικογενειών. Δεν πρόκειται για μομφή αυτό, δεν πρέπει κανείς να συμφωνεί απόλυτα με, την, ε, το πολιτικό του κόμμα. Εγώ στη διάρκεια της καριέρας μου πολύ συχνά διαφώνησα με το πολιτικό μου κόμμα. Αλλά όταν μιλάμε για συνοχή και συνεργασία ανάμεσα στα θεσμικά όργανα, εδώ είμαι πολύ επιτητικός και κάνω ό,τι μπορώ, ό,τι είναι δυνατόν για να υπάρξει συνεργασία. Θα έλεγα λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία σε κάθε πολιτικό επίπεδο ώστε οι αποφάσεις να είναι πιο συνεκτικές από, όσο είναι σήμερα. Συμφωνώ με αυτούς που λένε ότι υπάρχει πολιτική λιτότητας και ότι δεν θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την κρίση μόνο μέσω αυτής. Σωστά, σωστά. Αλλά είναι απαραίτητη αυτή η πολιτική αν ήμασταν παλαιότερα πιο προσεκτικοί και στο μακροοικονομικό επίπεδο και στο δημοσιονομικό επίπεδο, σήμερα δεν θα βρισκόμαστε στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Αλλά πράγματι χρειάζεται και μια θετική πολιτική ανάπτυξης και απασχόλησης. Και χαίρομαι παρά όλα τα αρνητικά στοιχεία που η ευρωπαϊκή οικονομία αναπτύσσεται μετά από περίπου 11 μήνες ύφεσης και το έχω, το έχω ξαναπεί ενώπιον αυτού του Κοινοβουλίου. Η κρίση της δεκαετίας του 30 ξεκίνησε από μια χρηματοοικονομική κρίση. Ποτέ δεν ελήφθη. Εμείς βρήκαμε θετική ανάπτυξη 11 μήνες μετά τη χρηματοοικονομική κρίση. Φέτος η μέση ανάπτυξη θα είναι περίπου το 1,5%. Κάποιες χώρες δεν έχουμε που δεν έχουν τα προβλήματα που γνωρίζουμε, θα υπάρχει ανάπτυξη του 2% και σε άλλες χώρες 3, ακόμα και 3,5%. Εν γέννη, για την στο επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αυξηθεί η απασχόληση. Φυσικά η ανεργία είναι υπερβολικά ψηλή. Χαίρομαι όμως γιατί σε σχέση με έξι μήνες νωρίτερα οι προβλέψεις μας για την ανάπτυξη είναι πολύ καλύτερες από ό,τι πιστεύαμε. Και επίσης η ανάπτυξη είναι πολύ πιο ισόρροπη από ό,τι πιστεύαμε. Δεν στηρίζεται μόνο στην αναπλήρωση ή στα διάφορα προγράμματα επανεκκίνησης ή στις εξαγωγές. Όχι. Είναι μια ανάπτυξη που επίσης τροφοδοτείται από την εσωτερική ζήτηση. Και στο τέλος θέλω να πω ότι παρά τα προβλήματα που γνωρίζουμε, οπωσδήποτε δε σε κάποιες χώρες, είμαι πεπισμένος ότι και πάλι θα νικήσουμε.